για την κατάσταση των δύο χριστιανών ιερέων στο Σουδάν. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους συντάκτες ε, των ψηφισμάτων αυτών. Η κυρία ε, Γιάννα Ζιτνάσκα έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η περίπτωση των δύο αυτών χριστιανών ιερέων με απασχολεί από την αρχή και μάλιστα είναι πάστορες οι άνθρωποι αυτοί και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Όπως γνωρίζετε, ε, συνελήφθη από τις μυστικές υπηρεσίες ο ένας ιερέας γιατί ε, είχε μιλήσει κατά της ε, αρπαγής γεών από το κράτος. Ο Μιχαήλ Γιάτη ήταν αυτός. Και μετά ε, ένας δεύτερος ιερέας που ε, ε, έψαξε να βρει τι έγινε, συνελήφθηκε αυτός και τους κατηγορούν για διάφορες κατηγορίες και κινδυνεύουν να τους επιβληθεί η θανατική ποινή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί μέσω της Αφρικανικής Ενώσεως να κάνει διαβήματα για να μην ε, εκτελεστεί η θανατική ποινή. Πριν από λίγες εβδομάδες ε, συνελήφθησαν 12 κορίτσια την ώρα που έβγαιναν από την εκκλησία. Και μάλιστα ε, ε τις μαστίγωσαν και όλα στη φυλακή της κοπέλες. Μπορεί κάποιος να αναρωτηθεί γιατί ασχολούμαστε με αυτά τα κράτη ε, που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα έχει νόημα πραγματικά. Ε, πέρυσι ε, λέγαμε ότι μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα για μια αντίστοιχη περίπτωση, περίπτωση ε, Ιμπραήμ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ζόρδη Σεμπαστιά. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου απευθύνατε το λόγο και στα Ισπανικά, μια γλώσσα που την αγαπώ και θα σας τα πω ε, και στα καταλανικά εγώ για, ε, όταν ε, μπορέσουμε βέβαια να έχουμε τη γλωσσική ισοτιμία εκφράζω την ικανοποίησή μου για το ψήφισμα και την ομοφωνία. Οι κρατήσει ε, ε, των δύο αυτών ε, παστόρων, Μάικλ Γιάτ και Γεν Ράιτ, είναι ακόμα μια εκτροπή τη κυβέρνηση του Σουδάν προ τον απολυταρχισμό. Είναι αυθαίρετε αυτέ οι καταγγελίες και ε, τιμωρούνται όπως ε, υπόθηκε πριν και με θάνατο. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι υπάρχει καταστολή, πρέπει να την καταγγείλουμε, πρέπει να καταγγείλουμε και τη θανατική ποινή ε, στο Σουδανικό Σύνταγμα, γιατί πολλοί εδώ πιστεύουν ότι με την θανατική ποινή κάτι μπορεί να λυθεί. Επίσης έχουμε την ριζοσπαστικοποίηση του καθεστώτος στην παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα υποστήριξης για τους δύο πάστορες, Ράιτ και Γιάτ, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι τους, ότι έχουν στο πλευρό τους την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πιστεύουμε στις αρχές της θρησκευτική ελευθερίας, δεν θα τους γυρίσουμε την πλάτη. Οι δηλώσεις αυτές όμως, αν δεν συνοδεύονται με οικονομική και πολιτική πίεση, δεν έχουν και πολύ αξία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και σας υπόσχομαι την άλλη φορά να σας τα πω καταλανικά. Στέτσινα. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα κύριε και κύριοι. Χαίρομαι που μαζί με άλλες πολιτικές ομάδες καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Και τώρα υποβάλλουμε ένα πολύ ισχυρό κείμενο που αποτυπώνει τη θέση μας και τη βούλησή μας να βοηθήσουμε τους ε, δύο ιερείς ε, που αντιμετωπίζουν ε, θανατική ποινή λόγω της χριστιανικής τους πίστης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τέκας που μου έδωσε τα κίνητρα για να συνταξώ το κείμενο αυτό τη δεκαετία του 90 όταν ε, οι χριστιανοί ε, του Νότιου Σουδάν έρχονταν ε, σε αντιπαράθεση με το Σουδάν ήταν μια εποχή πείνας όπου το Νότιο Σουδάν πάλευε για την ανεξαρτησία του και όπου οι Σουδανοί χρησιμοποίησαν σοβιετικά τάγκς ήταν μια εποχή όπου κάποιοι πουλούσαν ως σκλάβους τους χριστιανούς, μαύρους χριστιανούς. και ήταν αδύνατο να σταματήσουν τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, το Σουδάν. Αυτοί οι δύο χριστιανοί ιερείς είναι η κορυφή του παγόβουνου μόνο. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στετίνα. Και τώρα η κυρία Μαρή Κριστίν Βερσιά. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Το ψήφισμά μας κυρίως βασίζεται στην κατάσταση των δύο χριστιανών παστόρων και λυπάμαι γιατί θα μπορούσε να είναι ευκαιρία να διατρανώσουμε και πάλι πόσο ε, αποδοκιμάζουμε ε, το καθεστώς μετά τις ε, τελευταίες εκλογές. Ποτέ δεν ήταν το καθεστώς τόσο ενωμένο. Το είχαμε πει επανειλημμένα και εμείς στις 9 Ιουνίου που έγινε μια διάσκεψη και όπου ορισμένοι που είχαν υπογράψει την έκκληση του Σουδάν δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν. Ο Αμίν Μετανή που είναι πρόεδρος των Σουδανικών Οργανώσεων Κοινωνίας Πολιτών που ήταν στην καρδιά του ψηφίσματος που εγκρίναμε το περισμένο Δεκέμβριο και ένας άλλος πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου. Οι εκλογές ήταν οθευμένε. Ο κύριος Μπεσίρ πήρε πάρο, ε, πάνω από 94%. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ο κίνδυνος να καταδικαστούν σε θάνατο ο Μικαέλ Γιάτ και ο Πέτερ Γιάν Ράιτ είναι ένα μόνο θλιβερό παράδειγμα. Βεβαίως θα πρέπει οι αρχές του Σουδάν να σέβονται την αρχή της πίστης, της συνείδησης ε, και της σκέψης. Την ελευθερία να πιστεύεις ή να μην πιστεύεις, αλλά εκφράζεσαι και ελεύθερο παντού. Έτσι την Δευτέρα που μας πέρασε ένα ηγέτης της ε, αντιπολίτευσης ε, ε, καταδικάστηκε σε 20 μαστιγώματα και αμέσως εκτελέστηκε αυτή η ποινή έξω από το δικαστήριο, οποία ταπείνωση. Επίσης, ε, εκφεύγει του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου ο Μπασίρ, ταξιδεύει, πάει στη Νότια Αφρική ανενόχλητος σε μία σύνοδο και εξακολουθεί ο στρατός να βομβαρδίζει τους αμάχους. Η ανθρωπιστική βοήθεια έχει μπλοκαριστεί. Η κατάσταση των γυναικών, ανεξαρτήτως θρησκείας, είναι ικτρή. Όλα αυτά θα πρέπει εμείς να στιγματίζουμε και να καταγγέλουμε. Και λυπάμαι που και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπήκε σε διαδικασία διαπραγμάτευση με ένα τέτοιο καθεστώς για τη μετανάστευση. Δεν έχει τίποτα να περιμένει από το ονομά Αλ Μπεσίρ. Μόνο ένα διεθνέ πρόσωπο του προ... Ε, ε, ε, τίνουμε και ξέρει πολύ καλά να το εκμεταλλεύεται, ενώ είναι υπόδικος. Θα πρέπει και στο Σουδάν και στα αλλού να ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να εξαγάγουμε τα απαραίτητα συμπεράσματα πολιτικού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ιβαν Γιάκοφσιτς τώρα παρακαλώ. Σουδάνα. Ευχαριστώ. Οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι του Σουδάν αναμένουν φυσικά την υποστήριξή μας. Οι δύο ιερείς οι οποίοι ανετιολόγητα έχουν συλληφθεί ε, θα πρέπει να έχουν την υποστήριξή μας. Θα πρέπει να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα, διότι αυτή τη στιγμή το Σουδάν είναι μια χώρα όπου όχι μόνο υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν στη φλέκη, είναι μια χώρα χώρα όπου διάφορα σύμβολα καταστρέφονται, εκκλησίες, ε, απαγορεύεται η οικοδόμηση νέων εκκλησιών και το, καταστρέφεται και το ανθρώπινο πνεύμα, το δικαίωμα της ελεύθερης θρησκευτική πεποίθησης, ε, υπονομεύεται το δικαίωμα του να πιστεύει κανείς ό,τι θέλει. Και εγώ ανέκαθεν μαχήθηκα για την ελευθερία, ε, για τη θρησκευτική ελευθερία και καταδικάζω τα όσα λαμβάνουν χώρα στο Σουδάν και πιστεύω ότι είμαστε αρκετά δυνατοί για να βοηθήσουμε τους δύο ιερείς. Ευχαριστώ. Ο κύριος, Ο κύριος για ένα λεπτό ε, I don't see. Mr. Biden. Α, δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Καλώς τότε. Ακολουθούν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Το λόγο έχει ο κύριος Τόμας Τεχόφσκι για ένα λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, η υπόθεση των δύο παστόρων, χριστιανών παστόρων, οι οποίοι τώρα διώκονται στο Σουδάν, δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Τα τελευταία πέντε χρόνια, δυστυχώς, Πολλές ήταν οι περιπτώσεις ε, διώξεων χριστιανών στο Σουδάν. Κατοντάδες μετά το εμφύλιο πόλεμο έχουν δε και χιλιάδες εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Πρέπει να υποστηρίξουμε τους χριστιανούς στο Σουδάν. Είναι αδύνατο να ανεχθούμε μία μειονότητα, το 3% μόλις του πληθυσμού ε, παρόλα αυτά, ε, αλλά να μην έχει κανένα ε, δικαίωμα, να μην μπορεί να ασκήσει τη θρησκεία του αυτό το 3%. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση και όχι μόνο για τους δύο αυτούς πάστορες, αλλά για όλους τους χριστιανούς στο Σουδάν, οι οποίοι διώκονται. Τέλος, ε, επιτέλους πρέπει να αναλάβει δράση. Έχουμε τη Μύρια Μιμπραχήμ το 2014 τότε απέδωσε η βοήθεια του Κοινοβουλίου. Ελπίζω και σήμερα να αποδώσει. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Η κυρία Κέγγι. Έχετε ένα λεπτό, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι χριστιανοί, οι ιερείς Μέκλιγιατ και Πιτρή Ανδρέτ αυτή τη στιγμή πληρώνουν το τίμα και ενδεχομένως με τη ζωή τους της πρόσβασης σε ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, την ελευθερία θρησκείας, συνείδησης και πεποίθησης. Κατηγορούνται στη χώρα τους, στο Σουδάν, για τα χειρότερα εγκλήματα. Ε, υφίστανται εξευτελιστική μεταχείριση και μπορεί να καταδικαστούν σε θάνατο. Ζητάμε οι δύο ιερείς να αποφυλακιστούν άμεσα και ανεφόρον ώστε να σταματήσει οποιαδήποτε μορφή παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οποιαδήποτε δίωξη και εκφοβισμός ε, ενώπιον των χριστιανικών κοινοτήτων. Θα πρέπει να βγούμε από τη λογική της ενορχήστρωσης της θρησκείας για πολιτικές σκοπιμότητες. Δεν μπορούμε πια να ανεχτούμε καθεστώτα που παραβιάζουν την δεύτερη άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών με κατάφορη παραβίαση των διεθνών συνθήκων που έχουν επικυρωθεί και τα καθεστώτα τα οποία προβλέπουν θανατική ποινή θα πρέπει να την καταργήσουν εντελώς. Αυτός είναι ένα από τους βασικούς μας σκοπούς. Θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μας ε, για την κοινωνία των πολιτών στο Σουδάν, τους ανθρωπιστικούς οργανισμούς και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ευχαριστώ. E ε, Ευχαριστώ. Από την Ίσια, e Γκέρι και ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ε, Στη θέση 6 είναι το Σουδάν ε, ως προς τη δίωξη των χριστιανών, 80 φέτος. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι χριστιανός στο Σουδάν. Το βλέπουμε με τους δύο πάστορες και τη μοίρα τους, ο Μίχαλ Γιάτ και ο Πέτερ Φαράιτ. Είναι πολύ οδυνηρή η περίπτωση και πολύ εύγλωτη για τη δίωξη αυτή, τους διωγμούς που υφίστανται. Και ευτυχώ που καταφέραμε με του συναδέλφου τη πολιτική μου ομάδας να ξεκινήσουμε μια πρωτοβουλία για αυτό το ψήφισμα κατά των διωγμών των χριστιανών. Ιδιαίτερα για του δύο πάστορες ισχύει αυτό και για άλλου. Είναι περίπου 100 εκατομμύρια χριστιανοί που διώκονται ανά τον κόσμο. Η θρησκευτική ελευθερία είναι θεμελιώδε δικαίωμα και χαίρομαι που το ακούσαμε σήμερα επανειλημμένα. Εμεί που είμαστε η Ευρώπη των αξιών θα πρέπει παγκοσμίω να αγωνιστούμε για αυτέ τι αξίε. Δεν επιτρέπεται να αφήνουμε έτσι ε, να να διώκονται χριστιανοί, να το ανεχόμεθα, να κοιτάμε από την άλλη μεριά, επειδή οι άνθρωποι θέλουν ελεύθερα να ζήσουν την πίστη τους. Γι' αυτό ζητώ εξ ονόματος της ομάδας μου, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, εγερθείτε μαζί μας κατά της ε, ε, δίωξη και του διωγμών των χριστιανών. Να βοηθήσουμε τους δύο πάστορες αυτούς να ξαναβρούν την ελευθερία τους και όλοι οι διωκόμενοι χριστιανοί τη ζωή τους με ειρήνη και ισότητα και δικαιοσύνη. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σον Για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ ως μέλος του ΕΛΚΑ. Χριστιανοδημοκράτης με υπότιτλο. Είμαστε κατά των διακρίσεων ιδίως ε, κατά των χριστιανών. Είναι κάτι που μας ε, πληγώνει πολύ. Και ιδίως εδώ που έχουμε δύο χριστιανούς ε, πάστορες, τον Πέτερ Γιάν Ράιτ και τον Μάικλ Γιάτ, οι οποίοι συνελήφθησαν και ίσως ε, αντιμετωπίζουν ε, και τη θανατική ποινή μόνο και μόνο γιατί άσκησαν τη χριστιανική τους πίστη. Αυτό είναι αποτροπιαστικό και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε σίγουρα ώστε οι δύο αυτοί οι καταπληκτικοί άνθρωποι να απελευθερωθούν. Ιδίω εφόσον το Σουδάν έχει ε, επικυρώσει ε, τις σχετικές συμβάσεις ε, του ΟΗΕ και της Αφρικανικής Ένωσης. Παραβιάζει όμω ή παραγνωρίζει εντελώ τι διατάξει αυτών των συμβάσεων και θα πρέπει κάτι να κάνει η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Το στομότερο δυνατό Επίση, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε και την κατάσταση στον Ταρφούρ όπου αντίστοιχε είναι οι διακρίσει, όπου έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων εκτοπιστέντων και 4,5 εκατομμύρια ε, χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Άρα χρειάζεται το Σουδάν τη βοήθειά μας. Ευχαριστώ. Δέχεστε την μπλε κάρτα από τον κύριο Ζήκα Καφνεύσκη. Mr. Oh, Λάθος κατάλαβα, λέει ο πρόεδρος. Δεν θέλατε να στήσετε κάρτα. Περάσουμε λοιπόν στον επόμενο μιλητή, Γιούρε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι πάστορες αυτοί δεν είναι θύματα ε, πεφωτισμένων Ισλαμιστών, αλλά μιας κυβέρνησης, ε, της ε, μυσαλλοδοξίας της κυβέρνησης, που είναι και η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι για να δράσουμε. Βλέπουμε τι γίνεται μεταξύ μουσουλμάνων και χριστιανών τον 21ο αιώνα στην Ευρώπη. Μπορούμε να μιλάμε για τη μετανάστευση και την κλίμακα ε, τη μετανάστευση. Μπορούμε να μιλάμε για τον Ισλαμικό μουσουλμανικό πολιτισμό και βέβαια μπορούμε να τα λέμε και είναι και δικαίωμα και ευθύνη να το κάνουμε γιατί είμαστε και για τους άλλους υπεύθυνοι. Κανένα όμως ευρωπαϊκό κράτος δεν διώκει μουσουλμάνους για ό,τι λέγεται στατεμένοι ή για τις θρησκευτικέ τους ή ε, λατρευτικές τους συνήθειες. Εδώ μπορούν όλοι να εκφράζονται ελεύθερα, να μιλούν για τις ε, προσδοκίες τους, για τα προβλήματά τους. Και είμαστε πάντα έτοιμοι να έχουμε διάλογο, να απαντήσουμε. Άρα έχουμε το να ζητήσουμε την ίδια αντιμετώπιση για τους χριστιανούς σε όλες τις μουσουλμανικές χώρες. Δηλαδή να αντιμετωπίζονται όπως αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ τους μουσουλμάνους. Βέβαια για να γίνει αυτό θα πρέπει να ταυτιστούμε με τους αδελφούς μας αυτούς γιατί πολλές φορές απειλείτονται και υποφέρει περισσότερο λόγω και της δικής μας αδιαφορίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Γιούρακ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτροπέ, η δυσαρεστή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συζητείται συχνά εδώ. Δεν θα επανελάβω τις διαφορές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν κάποιες ε, ακτίδες ελπίδας. Πριν από ένα χρόνο, σύντομα, αμέσως μετά από την έγκριση του ψηφίσματός μας, η Μίρια Μιμπραχήμ, μια χριστιανή που καταδικάστηκε θα, είχε καταδικαστεί σε θάνατο, αποφυλακίστηκε. Οπότε οι προσπάθειε δεν είναι Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να θυμάται το σύσταση του Συμβουλίου του 2013 όπου λέγεται ότι θα προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια αλλά υπό τον όρο ότι ε, τηρείται η ελευθερία ε, θρησκείας. Μπορούμε λοιπόν πιστεύω και με αυτές τις προσπάθειες που έχουμε τώρα και αυτό το ψήφισμα να έχουμε την ίδια επιτυχία όπως πριν από ένα χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στο Κατσδιάι. Ανάζα Μπόλσκα. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όταν μια χώρα κατηγορεί δύο χριστιανούς πάστορες ότι έχουν κηρύξει τον πόλεμο στη χώρα, καταλαβαίνετε περί τίνος πρόκειται. Ότι είναι ψευδής η κατηγορία. Ο πόλεμος ε, το Ισλάμ κατά των χριστιανών αρχίζει όταν αρχίζουν να καταδαφίζουν εκκλησίες οι ίδιοι. Και όταν δεν γίνονται σεβαστά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και το ελάχιστο που μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να καλέσουμε τις κυβερνήσεις και τη συγκεκριμένη κυβέρνηση ε, να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει εκεί. Αυτό το οφείλουμε στους συντάκτες ε, των ψηφισμάτων. Θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οποία αλαζονία. Μιλάμε για τη δίωξη των χριστιανών στο Σουδάν και πριν από τρεις ώρες στην έκθεση της γειτονίας ε, δεν ε, ψηφίσαμε υπέρ των διωγμών των χριστιανών. Το βγάλαμε από το ψήφισμα. Εν πάση περιπτώσει. Ο πρόεδρος, η κυρία Άννα Γκόμες, παρακαλώ θα ήθελα να πω ότι το 2004 είχα πάει στο Σουδάν και στο Ταρφούρ το 2010 και το 2011 ως ε, μέλος του Κοινοβουλίου για την παρατήρηση των εκλογών. Και είδαμε πώς είχε τότε η κατάσταση. Τότε η ε, κυβέρνηση του Ομάρ Αλμπασίρ ε, εδίωκε τους χριστιανούς ήδη από τότε όπως και τους δύο πάστορες που έχει φυλακίσει τώρα και κινδυνεύουν να χάσουν και τη ζωή τους ε, πέρα από τα βασανιστήρια. Η χώρα αυτή ε, ε, καταπιέζει το λαό του με τρομερή καταστολή, βία. Θα πρέπει να το καταλάβει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δίκες είναι εικονικές, είναι Η κυβέρνηση στρέφεται κατά του λαού της και παράγει μετανάστες. Δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ο τελευταίος προστάτης του Μάραλ Μπασίρ και να σταματήσει η διαδικασία του χαρτούμ για τη μετανάστευση. Είναι φυγόδικος, το ψάχνει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Θα πρέπει εμείς να μιλάμε και να είμαστε φωνή των θυμάτων αυτού του καθεστώτος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους συντάκτες αυτής της ε, πρότασης ψηφίσματος, λέει και ο ε, Κρασνοντεύσκη. Θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά πώς έχει η κατάσταση των χριστιανών στις μουσουλμανικές χώρες. Αυτό το λέει και η ομάδα μου και το υποστηρίζει συχνά. Θα ήθελα εδώ να εκφράσω ένα φόβο όμως μήπως πρέπει να έχουμε ε, άλλου είδους συζητήσεις εδώ, σε άλλο ύφος και σε άλλο τόνο. Τι σπταίει για την αδιαφορία αυτή ε, για των πεπρωμένων και τη ζωή των χριστιανών που διώκονται σε πολλά μέρη του κόσμου. Γιατί καμιά φορά βλέπω αντιστάσεις εδώ κατά της αναγνώρισης ε, και κατά της διαπίστωσης κάνω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα περιθωριοποιούνται οι χριστιανοί στην Ευρώπη και στη δημόσια ζωή. Άρνοτ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, η έκθεση αυτή δεν είναι τέλεια, αλλά η αρχή βρίσκεται μέσα. Σύμφωνο με τους υπόλοιπους εδώ, λέγοντας ότι η θανετική ποινή για τους ε, χριστιανούς οπουδήποτε στον κόσμο είναι κάτι απολύτως απαράδεκτο. Ξέρετε ότι εγώ είμαι μέλος του UKIP στο Κοινοβούλιο και είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε τα επόμενα μου λόγια μπορεί να σας κάνουν εντύπωση. Αλλά εγώ θα ψηφίσω υπέρ αυτού του ψηφίσματος και παρατρενώ ολόκληρη την ε, αίθουσα εδώ, ολόκληρο το Κοινοβούλιο να κάνει το ίδιο. Ευχαριστώ. Λοιπόν τώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η κυρία Επίτροπο Σεσίλια Μάλμστρομ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε είναι καλή ευκαιρία να που κάνουμε αυτή τη συζήτηση με εμένα εδώ εκ μέρους της ε, είπα της εκπροσώπου για τις ε, δύο δίκες των δύο ιερέων που αναφέραμε σήμερα στο Σουδάν και οι δύο ιερείς αυτοί ανήκουν στην Ευαγγελική Πρεσβυταριανή Εκκλησία στο Χαρτούν και αυτή η εκκλησία ε, κατεδαφίστηκε από τις ε, Εθνικές Υπηρεσίες Πληροφοριών του Σουδάν ε, ε, κατηγορούνται για υπονόμωση του συνταγματικού συστήματος και για κατασκοπία που όπως αναφέρατε μπορεί να οδηγήσει τη θανατική ποινή. Η προανάκριση τελείωσε 7 Ιουλίου και ελπίζουμε να έχουμε κάποια καλά νέα. Ειδικότερα διότι τα αποδεικτικά στοιχεία δεν ήταν βάσιμα. Δυστυχώ ο δικαστή αποφάσισε να δεχθεί την υπόθεση και θα γίνει κανονικότατα η δίκη στι 14 Ιουλίου. Και να είστε βέβαιοι ότι θα την ακολουθούμε στενά. Η αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο Χαρτούμ ε, ήταν σε στενή επαφή με του δικηγόρου των ιερέων σε όλη τη διάρκεια τη υπόθεση και ε, τους παρέχουν συμβουλή για τις προνακρίσεις θεωρούμε ότι αυτό στέλνει ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα για το πόσο σημαντική είναι για μας η διαδικασία και ειδικότερα η ελευθερία της θρησκείας, της ε, πίστης, ε, της έκφρασης και του δικαιώματος για δική δίκη. Αυτό απεικονίζει για άλλη μια φορά την βαθιά ανησυχητική κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των θεμελιδών ελευθεριών γενικότερα στο Σουδάν καθώς ε, και την μέγενη που των κρατικών δυνάμεων στα κρατικά ιδρύματα ειδικότερα ε, όπως βλέπετε την κατάσταση των Ταρφούρ ε, και σε άλλα μέρη ε, που οδηγεί πάρα πολλούς ανθρώπους στη δυστυχία. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιμείνουμε για την απελευθέρωση των δύο ιερέων και για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με όλους τους ενδιαφερομένους του Σουδάν. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Έχω λάβει έξι σχέδια ψηφισμάτων από διάφορες πολιτικές ομάδες. Οπότε κλείνουμε αυτή τη συζήτηση και θα ψηφίσουμε τώρα για